προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Ο εισηγητής έχει τέσσερα λεπτά για την εισαγωγή της εκθεσής του. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την έκθεση αυτή πρέπει να κατανοήσουμε την πολιτιστική σπουδαιότητα της πολιτισμικής κληρονομιάς και τις ευκαιρίες που ε, ενέχονται εδώ για τις ε, κοινότητες και τους πολίτες είναι μια ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση αναφέρεται και στον τίτλο ολοκληρωμένη σφαιρική σημαίνει ότι στην πρακτική εφαρμογή θα πρέπει να είμαστε ε, στην προσέγγιση μας στην καθημερινή μας δράση να λαμβάνουμε υπόψη αυτή τη διάσταση κάποια σημεία θα ήθελα να τονίσω για να ε, ξεκινήσω και το ευρωπαϊκό έτος της πολιτισμικής κληρονομιάς ε, με τον εξοπλισμό, την πρικοδότηση από πλευράς κονδυλίων από τον προϋπολογισμό με τις καλύτερες πληροφορίες ε, για την ε, προώθηση της πολιτισμικής κληρονομιάς με μια ενιαία θηρίδα για τις δράσεις αυτές. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι η πολιτισμική κληρονομιά απαιτεί πάρα πολλούς επενδυτές και επιχειρηματίες στα πολιτισμικά θέματα που πρέπει να έχουν δυνατότητα να δρουν μέσα σε ένα σφαιρικό πλαίσιο. Και από το ΦΕΝΤΕΡ και τα κονδύλια τα οποία διαθέτουμε για τον πολιτισμικό τομέα κάνουμε πραγματικά, ε, δίνουμε αγώνα για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτά τα κονδύλια και αυτές τις δυνατότητες. Και πρέπει εδώ σε σχέση με τους πολίτες ε, να υπάρξει η δυνατότητα να συνεισφέρουν και από πλευρά τους να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια. Ένα άλλο θέμα είναι ο έλεγχος των σχεδίων και των προγραμμάτων για την πολιτισμική κληρονομιά. Δεν είναι μόνο μια απαρίθμηση παραγόνων και συνιστών είναι μια σφαιρική δράση που πρέπει να οδηγεί στο να δημιουργούμε χειροπιαστά και να συμπεριλαμβάνονται μια ολόκληρη σειρά μέτρων με την ε, αναφορά στην ποιότητα και την αναβαθμισμένη ποιότητα σε σχέση με το έργο που πρέπει να αναπτύξουμε όσον αφορά τα πολιτισμικά θέματα. Επίσης πρέπει να υπενθυμίσουμε κάτι εδώ, το ότι η ε, επίθεση η οποία έγινε στην Παλμύρα από το Ίκη στο Ισλαμικό κράτος Ιράκ και Συρίας με την καταστροφή ναών στην Παλμύρα που ήταν πραγματική ε, παγκόσμια κληρονομιά όπως είχε χαρακτηριστεί ε, από την UNESCO παγκόσμια κληρονομιά σε αυτό το μνημείο είναι εγκληματίες αυτοί οι οποίοι διέπραξαν αυτό το έγκλημα καταστρέφοντας αυτό το ναό ε, καταστρέφοντας έτσι ένα μνημείο της πολιτισμικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Και αναφέρομαι εδώ σε σχέση ε, με προτάσεις που έγιναν για να μπορέσουμε να ε, έχουμε την ε, διάχυση των δράσεών μας για την διασφάλιση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Πρέπει να σας πληροφορήσω ότι η πρόσφατη αξιολόγηση όσον αφορά τις ζώνες κινδύνου ε, σε σχέση και με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση η αξιολόγηση αυτή όσον αφορά και γεωπολιτικά κριτήρια και στρατιωτικά και οικονομικά κριτήρια τα οποία όλα εμπλέκονται σε σχέση ε, με τις υποθέσεις αυτές και όχι μόνο αποκλειστικά πολιτισμικά κριτήρια αποκαλούμενη κρίση των προσφύγων όπως την αποκαλούμε σήμερα, το προσφυγικό δηλαδή ζήτημα με τις ε, τεράστιες μεταναστευτικές ροές που έχουν προκληθεί, εδώ ενέχεται ο κίνδυνος να ε, υποκρύπτεται μια άλλη κρίση η οποία υποβόσκει και είναι πολιτισμικού χαρακτήρα. Εδώ αγνοούνται και καταστρέφονται πολιτισμοί από την, ε, που αποτελούν κληρονομιά της ανθρωπότητας. Κύριε Κρυστοφόρη, το λόγο για ένα λεπτό. Για μένα η Ευρώπη είναι ο ορισμός του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και θεωρώ ότι η Ευρώπη έπρεπε να είναι και να παραμένει θεματοφύλακας ολόκληρης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Προέρχομαι από μια χώρα την Κύπρο που εδώ και 41 χρόνια ανεκτήμητης και αμύθιτης αξίας, πολιτιστική και θρησκευτική θησαυρή, λαιλατήθηκαν, συλλήθηκαν και αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στο λαθρεμπόριο, στα χέρια των λαθρεμπόρων, ακόμα και μέσα στην Ευρώπη. Η Κύπρος είναι μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς. Δικαίως αποκαλείται ότι είναι η νήσος των Αγίων χιλιάδες εκκλησίες χιλιάδες μνημεία χιλιάδες χρόνια πολιτισμού θρησκευτικού και αρχαιοτήτων καταστράφηκαν και εμπορεύονται αυτή τη στιγμή ακόμα και μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Όταν κλέβεις μια αρχαιότητα από ένα μουσείο είναι έγκλημα. Όταν καταστρέφεις πολιτιστικά μια χώρα για μένα είναι έγκλημα καθοσιώσεως. Αναμένω από την Επιτροπή στην οποία αναπευθύνθηκα πολλές φορές όχι μόνο να πάρει μέτρα αλλά να θεσπίσει νομοθετικό πλαίσιο για αυτόματον επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων που διακινούνται στην Ευρώπη για να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για να υπάρξουν χώρε, όπω είναι η Κύπρο αλλά και άλλε χώρε όπω αναφέρθηκε προηγουμένω η Παλμύρα στη Συρία και σε άλλε περιοχέ του κόσμου. Σα ευχαριστούμε πολύ, αλλά στηρίσουμε το χρόνο αγόρευση. Η κυρία Κώστα έχει το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Διάκονο για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Πραγματικά εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά με ένα πολύ ουσιώδε ζήτημα, την πολιτιστική κληρονομιά και θελήσαμε μέσω τη έκθεση αυτή να δώσουμε συνέχεια στην ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να έχουμε και μια έκθεση όμω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα ζητά από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουν τη δέσμευσή του όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Αποτελεί άξονα ανάπτυξη η πολιτιστική κληρονομιά, αποτελεί άξονα απασχόληση, αποτελεί άξονα επέμβαση όσον αφορά ακόμα και τι επενδύσει και είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει μια έντονη συμβολική σημασία για την πολιτιστική κληρονομιά. Βέβαια έχουμε κάποια τραγικά γεγονότα τα οποία μας τα υπενθύμησε και ο εισαγητής. Ξέρετε ότι στις 15 Σεπτεμβρίου θα γιορτάσουμε την επέτειο της ε, Σύμβασης Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε τι μας ζητάει η έκθεση αυτή. Να έχουμε καταρχάς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση οριζόντια για όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομία και να κινητοποιηθούν όλοι οι φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελεί τεράστια περιουσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, με αφορμή τη συζήτηση για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης θα ήθελα να ενημερώσω για άλλη μια φορά το σώμα ότι κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής λαιλάτισαν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της πατρίδος μου της ελλάδας. μάλιστα η λίστα με τους κλαπέντες αρχαιολογικούς θησαυρούς περιέχεται τόσο στον ειδικό τόμο που εξέδωσε το 1946 το ελληνικό υπουργείο παιδείας όσο και στην αντίστοιχη ειδική έκθεση που συνέταξε το βρετανικό υπουργείο πολέμου σύμφωνα με την οδηγία ενενήντα τρία 7 ΕΟΚ που αφορά στην επιστροφή στον τόπο προέλευσής τους των κλαπέντων αρχαιολογικών θησαυρών αλλά και τη σύμβαση unesco unidroit του 1970 προβλέπεται ο επαναπατρισμός των πολιτιστικών αγαθών. επομένως κύριε επίτροπε σας επαναφέρω το θέμα το οποίο σας έθεσα και την ημέρα πριν ένα χρόνο όταν γινόταν η συζήτηση προκειμένου να είστε υποψήφιος επίτροπος και σας είχα θέσει το θέμα αυτό. έχετε μια απάντηση για την επιστροφή των κλαπέντων αρχαιολογικών θησαυρών από τους ναζί την επιστροφή τους στην ελλάδα. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Γιάκοβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι ε, η Αμερική θα γίνει ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο, η Ασία ένα τεράστιο εργοστάσιο και η Ευρώπη τελικά θα παραμείνει ένα μουσείο. Αυτό λένε πολλοί. Σε 100 χρόνια λένε ότι έτσι θα διαμορφωθούν τα πράγματα στον κόσμο. Και κατά αυτόν τον τρόπο τελικά είναι σαν μας λένε ότι η ηλική και άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω το ακόλουθο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι σημαίνει ο πολιτισμός για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Μόνο και μόνο αυτό αξίζει να εξετάσει κανείς και θα καταλάβει τη διάσταση του ζητήματος. Πόσο σημαντική είναι η πολιτιστική κληρονομιά για την ταυτότητά μας αλλά και για την οικονομία μας. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω το σχέδιο των ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτευουσών, αλλά παράλληλα με τέτοια προγράμματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ενδεχομένως να θεσπίσει και συγκεκριμένε περιφέρειες ως πολιτιστικές περιφέρειες Ευρώπης, όχι μόνο τις πρωτεύουσε. Ο κύριος Μάραγκαλ έχει το λόγο. Για την καταστροφή της Παλμύρας είναι ένα τρομερό παράδοξο, ένας, ένας παραλογισμός. Τουλάχιστον ελπίζουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να συνειδητοποιήσει περί τίνος πρόκειται. Είναι ρητή η ε, τοποθέτηση του τίτλου ε, towards ε, δηλαδή προς μια συνεκτική πολιτική στην Ευρώπη με δράσεις ε, στρατηγικές με δυνατότητα διασφάλισης αυτών των συνιστοσών. Να το πούμε ξεκάθαρα που μας λέει αυτή η έκθεση αν θέλουμε να διασφαλιστεί και να σωθεί η Ευρώπη μελλοντικά πρέπει να σωθούμε την, να γνωρίσουμε και να αξιολογήσουμε και να σεβαστούμε την ιστορία μας που πάντα είναι εκείνο που συνοδεύει την θρησκευτική, οικονομική και άλλη δράση σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε μια συγκεκριμένη πολιτισμική ενότητα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια οδό με σωστέ προθέσεις. Ζητείτε λοιπόν μια ενιαία θηρίδα στην Ευρώπη που θα συντονίζει τις διάφορες δράσεις στην Ευρώπη και ταυτόχρονα θα αναγνωρίζει τις περιφέρειες και πόλεις που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής στην Ευρώπη. Ευχαριστώ.

αξιότιμοι ευρωβουλευτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να ευχαριστήσει τον εισηγητή κύριο Διακόνου και τους σκιώδεις εισηγητές για την ποιότητα και το θετικό πλαίσιο της έκθεσης. Καλύπτεται το σύνολο του εύρους της πολιτιστικής κληρονομιάς με προτάσεις και συστάσεις και βήματα και διαβήματα που πρέπει να αναλυφθούν. Σημερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψη του ότι υποστηρίζοντας και ενδυναμώνοντας την πολιτισμική διάσταση για την πολιτιστική κληρονομιά έχει τεράστια σπουδαιότητα. Η πολιτιστική κληρονομιά συνεισφέρει σημαντικά και στην οικονομική και στην οικονομική ανάπτυξη. Αφορά τη ζωή όλων των Ευρωπαίων και αφορά το αίσθημα που έχουν ότι ανήκουν και έχουν ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μιλώντας αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι γίνονται πράξεις βανδαλισμού που καταστρέφουν μνημεία όπως βλέπουμε με τις εικόνες καταστροφής μνημείων στο Ιράκ και στη Συρία. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα όσον αφορά την πολιτισμική κληρονομιά. Ε, η χρήση του ιστορικού αυτού πλαισίου πρέπει πραγματικά να μας κάνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τη διασφάλισή του. Πρέπει να εξευρεθούν τα σωστά μέσα και μέτρα για να επιτευχθεί πρόοδος στην αναζήτηση μηχανισμού πολιτισμών και πολιτικών και στρατηγικών για την ένταξη αυτών των συνιστοσών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ήδη έχει αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολλά από αυτά τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση. Έχει ξεκινήσει να συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη σε ένα συμμετοχικό πλαίσιο. Το 2016, το 2017 θα συνεχιστεί αυτό το έργο για την κατάρτιση, εκπαίδευση και διάχυση γνώσεων. Επίσης οι γνώσεις διαδίδονται μέσω των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της πόλης με τις βέλτιστες πρακτικές και τις καλύτερες δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να διευρύνει την εσωτερική συνεργασία και τη διαθεσιμότητα δυνατοτήτων και δράσεων ώστε να μπορούν να ευδοκιμήσουν μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και εδώ θα ήθελα σε σχέση με τις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών να πω δυστυχώς η απάντησή μου είναι η ίδια όπως και κατά την ακρόαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εξουσίες ε, για την ε, αντιμετώπιση θεμάτων όσον αφορά διαφορετικά κράτη-μέλη. Αυτά είναι θέματα διμερών διαφορών που πρέπει να επιλύονται μεταξύ των κρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συζήτηση και θα ψηφίσουμε